Shall I start again? I think the problem is that... Πρόεδρε, το πρόβλημα είναι ότι εμ, έκανε ένα reset όλο ο, ο εξοπλισμό εξοπλισμός ε, και ενδεχομένω κάποιοι να μην το αντιλήφθηκαν. Αλλά επανεκκινήθηκαν όλε τι κονσόλε εδώ τη Γερμανίας. I don't mind starting again, if that, if that helps πρόσωπο της Επιτροπής. Ε, καλώς να ξεκινήσω και πάλι από την αρχή. Ελπίζω να μπορείτε να με ακούσετε όλοι. Λοιπόν, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, ξεκίνησαν μια διαδικασια αντι anti-dumping και αθέμη των ενισχύσεων σε ό,τι αφορά επιτραπέζιες ελιές προέλευση Ισπανίας στις 13 Ιουλίου του 2017 οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, προφανώ έχουν το δικαίωμα να ξεκινήσουν μια τέτοια ε, έρευνα στο πλαίσιο του ΠΟΕ, αλλά δεν αποτελεί μυστικό ότι μα ανησυχεί πολύ εν λόγω έρευνα. Και ποιο είναι ο βασικό λόγο, όχι μόνο επειδή μα ανησυχούν οι δυνητικέ ανδικέ συνέπειε που αυτό θα μπορούσε να έχει για του παραγωγού τη πανητή ελιά, αλλά και επειδή θεωρούμε πω τα καθεστώτα ενίσχυση τα οποία υποτίθεται πως εντόπισε οι Ηνωμένες, ε, Πολιτείες ε, ε, δεν προβλέπουν σε, ή μάλλον δεν δημιουργούν στρεβλώσεις στο εμπόριο. Δηλαδή περιλαμβάνονται στις επιτροπόμενες ενισχύσεις. Οπότε μας ανησυχούν οι δυνητικοί συστημικοί, δυνητικές συστημικές συνέπειες που θα μπορούσε να είχε λήψει τέτοιου είδους μέτρων. Τώρα, από την αυτή εξ αρχή, ε, από την αρχή αυτή τη διαδικασία, εμεί συνεργαστήκαμε από την πλευρά τη Επιτροπή, δηλαδή με τι ε, Ισπανικέ Αρχέ και τι σχετικέ ε, επιχειρήσει, προκειμένου να αντιταχθούμε και ήδη έχουμε απευθυνθεί και γραπτό και προφορικό στην αρμόδια για αυτήν την έρευνα αρχή των Ηνωμένων και προφανώ βρισκόμαστε στη διάθεσή του ε, για να παράσχουμε στην Ισπανική κυβέρνηση και στου ε, παραγωγού ε, τη Αλιάς τη Ισπανίας οποιαδήποτε υποστήριξη. Ακριβώ επειδή μα ανησυχεί ο δυνητικό συστημικό διεκτυπώ, έχουμε σε υψηλό πολιτικό επίπεδο έχουν υπάρξει επιστολές από του επιτρόπου Χόγκαντε Μάστρομ αλλά και από την πλευρά ε, της ε, αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, οι γραμματείς δηλαδή Ποντιού και Ρος, οι οποίοι με επιστολή τους εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία σε ό,τι αφορά αυτά τα μέτρα και υποστηρίζουν ότι δεν είναι προς το συμφέρον των ίδιων των Ηνωμένων πολιτιών να εφαρμόσουν ε, μέτρα ε, κατά των ενισχύσεων σε ό,τι αφορά ενισχύσεις οι οποίες δεν, έχουν, ε, δεν δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά. Αναμένουμε τώρα τις, τα προκαταρκτικά απορίσματα σε ό,τι αφορά αυτές τις αθέμητες, υποθέμενες ασέμενες ενισχύσεις και τα μέτρα αντι-dumping προς τα τέλη του Νοεμβρίου και από εκεί και μετά θα υπάρξουν και κάποιε επισκέψει επαλήθευση, από το Υπουργείο δηλαδή Εμπορίου ε, στους ε, παραγωγούς ε, τη Ισπανία. Και εμεί βέβαια θα παρευρεθούμε από την πλευρά τη Επιτροπή προκειμένου να υποστηρίξουμε του παραγωγού σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα που θα του τεθούν και μόνο το Φεβρουάριο του 2018 θα υπάρξει το τελικό πόρισμα σε ό,τι αφορά αυτές τις υποτιθέμενες αθέμητες ενισχύσεις και, τα, το υποτίμηνο ντάμπινγκ. Και μόνο μέσα στο Μάρτιο θα υπάρξει τελικά η τελική απόφαση που θα ληφθεί και ενδεχομένω τελικά, η οποία ενδεχομένω να οδηγήσει στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Για παράδειγμα, επιβολή επιπρόσθετων δασμών ε, σε ό,τι αφορά τι συγκεκριμένε ελιέ και την εισαγωγή του στι ΗΠΑ. Είναι λίγο πρόημο το να υποθέτουμε ω προ το ποιο θα είναι το τελικό πόρισμα. Ελπίζουμε δηλαδή ότι το ε, Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα λάβει υπόψη τα σχόλια μα και θα καταλήξει σε ένα πόρισμα που δεν θα οδηγήσει στην επιβολή συμπληρωματικών δασμών, αλλά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά ε, τι εξελίξεις και θα δούμε εάν θα χρειαστεί στο μέλλον να λάβουμε και εμεί συμπληρωματικά μέτρα από την πλευρά μα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πριν συνεχίσουμε να καλωσορίσω εκπροσώπους από το κλάδο παραγωγής ελαιών στην Ισπανία με πρόσκληση των Ισπανών Ευρωβουλευτών. Τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, επόμενο καλεσμένο μας εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διάθεση Γεωργίας. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά σε αυτά που είπε ο κύριος Ρουμπινάτσι που μίλησε για τα για τους μηχανισμούς προστασίας του εμπορίου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και μας προβληματίζει και ανισχύει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ε, στρέφεται, στρέφονται οι Ηνωμένε Πολιτείε κατά επιδοτήσεων της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, που δεν αφορούν συγκεκριμένο προϊόν ούτε στρεβλώνουν τον ε, ανταγωνισμό και μάλιστα προειδοποίησαμε τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές. Στείλαμε ένα μήνυμα με τις ανησυχίες μας και είπαν ούτως ή άλλω με βάση το Green Box του ΠΟΕ και οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν αντίστοιχε επιχορηγήσει. Ε, στα τέλη του επόμενου θα έχουμε την Υπουργική Διάσκεψη των Buenos Aires στα πλαίσια του γύρου του διαπραγματεύσεων τη Ντόχα. Εκεί θα γίνουν πολύ κρίσιμες συζητήσει. Ε, οπότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλα τα μέλη του ΠΟΕ για μεταρρύθμιση των ε, ε, συστημάτων γεωργικών επιδοτήσεων. Είναι μια συζήτηση που διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια και μια και οι ΗΠΑ μέχρι στιγμή ήταν σημαντικό μα εταίρο ε, και συμβαδίζαμε ε, σε πολλά θέματα. Και μάλιστα ε, είπαμε ότι θα μεταβούμε σε ένα σύστημα επιδοτήσεων που δεν θα είναι στρεβλωτικό για τον ανταγωνισμό. Σε επιδοτήσεις τύπου green box, κάτι που κάναμε στο παρελθόν, επιδοτήσεις διαστρέβλωναν τον ανταγωνισμό. Πάντως ε, θα έχουμε συνεργασία και συντονισμό και με τους ενδιαφερομένους. Είναι πολύ επώδυνη αυτή η διαδικασία της ε, έρευνας. Ουσιαστικά στέλνουν ερωτηματολόγια 200 σελίδων σε όλες τις αρμόδιες αρχές της Ισπανίας, ε, ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς προσπαθούμε να συντονίσουμε τις απαντήσεις στα μεμονωμένα ερωτηματολόγια, είτε απευθύνονται στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα της Μαδρίτης, είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπως είπε ο κύριος Ρουμπινάτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει το παρόν και είναι στη διάθεσή σας για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας. Μπορούμε μάλιστα και επιτόπου να μεταβούμε ε, σε έρευνες ε, όταν θα στείλουν τα κλιμάκια τους οι Ηνωμένε Πολιτείε στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία για να πραγματοποιήσουν τις έρευνες. Μπορούμε να είμαστε και εκεί παρόντες. Ευχαριστώ κυρία Εράς Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το, την υψηλή εμπλοκή της ε, στο θέμα αυτό, γιατί είναι γεγονός ότι ε, ε, εξ αρχής ξεκίνησαν σε συνεργασία με την Ισπανική κυβέρνηση να συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο προέκυψε μετά από την ε, ε, προώθηση ε, από πλευρά της Κομισιόν ενός προγράμματος για τη βελτιστοποίηση της προώθησης της Ισπανικής ελιάς στην Αμερικανική αγορά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης ότι εδώ και πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τροποποιήσει τις ενισχύσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής έτσι ώστε να Στρεβλώσει στρεβλώσεις ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο, ότι οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν η παραγωγή ελιάς είναι στο green box, δεν προκαλούν καμία απολύτως στρέβλωση στην ε, διεθνή αγορά και επομένως εδώ δεν μιλάμε για την προστασία ε, των ε, παραγωγών ελιάς μιας συγκεκριμένης χώρας, αλλά να υπεραμεινθούμε της κοινή γεωργικής πολιτικής απέναντι σε επιθέσεις από πλευράς παραγωγών ε, της Βόρειας Αμερικής. Ε, νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι σαφές ε, ότι οι δικές μας ενισχύσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις τρευλωτικές πραγματικά πρακτικές στήριξης εισοδήματος κλπ. που ισχύουν στην Βόρεια Αμερική. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε όμοιροι στον τομέα της επιτραπέζης τραπέζιας βρώσιμης ελιάς. Αλλά αύριο μπορεί να είναι ένας άλλος τομέας. Ε, και νομίζω ότι ε, με αυτόν τον τρόπο ε, η κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ προσπαθεί να επιτεθεί στην κοινή γεωργική μας πολιτική και τις πρακτικές μας. Ευχαριστούμε πολύ του, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν εμπλεκεί και συνεχίζουν να ε, ε, υπεραμείνονται ε, της ελιάς αλλά και της ιωικής πολιτικής γιατί οποιασδήποτε επιδοτήσεις υποστήριξης εισοδήματος εμπίπτουν στο Green Box δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα όσον αφορά τον όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την Κομισιόν, να ευχαριστήσω την Ισπανική κυβέρνηση για την εργασία που έχουν κάνει και θα συνεχίσουν να κάνουν τους επόμενους μήνες και να υπενθυμίσω ότι τελικά όμοιροι κρατούνται η παραγωγή της ελιάς αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Λουαζό. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε της παντοδύναμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Αμερικανικές αρχές ε, θέλουν να επιβάλλουν μέτρα αντι-dumping απέναντι στις εισαγωγές ελιάς από την Ισπανία. Θεωρούν, είπα, ότι οι τιμές της Ισπανίας είναι dumping λόγω των επιδοτήσεων των ελιών της ε, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την τον Αμερικανικό κλάδο, γιατί και οι Αμερικανοί ε, παράγουν ελιές, στην Καλιφόρνια κυρίως. Εγώ είμαι υπέρμαχος του προστατευτισμού και πραγματικά όχι μόνο κατανοώ, αλλά και επικροτώ αυτή τη βούληση των Αμερικανών να προστατεύσουν τα προϊόντα του, αλλά αντιλαμβάνομαι και την ε, αίσθηση της ανυμπορίας που νιώθουν οι ε, ισπανή παραγωγή απέναντι σε αυτή τη στάση των Αμερικανών. Τι μέτρα θα λάβει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν επιβεβαιωθεί η βούληση των ΗΠΑ να προστατεύσει τα προϊόντα της. Επίσης, ε, τι ε, δράση θα αναλάβουμε ε, απέναντι στου Αμερικανούς που προτάσουν τα συμφέροντα των παραγωγών τους. Περάνω πάντω άλλου πράγματο. Και Μήπως θα πρέπει να επιβάλλουμε οικονομικά αντίκτυπα σε περίπτωση εφαρμογής τέτοιες προστατευτικής πολιτικής από τη ΣΥΠΑ. Ε, καταλαβαίνω τη θέση σας που πραγματικά φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολη και περιμένω απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που προβλέψαμε τη συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή μας, γιατί είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί και προβληματίζει τους Ισπανούς ελαιοπαραγωγούς, αλλά όχι μόνο γιατί πρόκειται για ένα πρόβλημα που μπορεί να αγγίξει την ίδια την ΚΑΠ και γι' αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μέχρι σήμερα. Και χαιρετίζω τους εκπροσώπους της Διαπαγγελματικής Οργάνωση Επιτραπέζιων Ελιών που ήρθαν και μήνες ολόκληρους ασχολούνται με το θέμα αυτό εκπροσωπώντας και προασπίζοντας τις ενισχύσεις της ΚΑΠ, όπως τα μέτρα περί οικολογικοποίησης, τα μέτρα του greening. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και 40 χρόνια εξάγουμε επιτραπέζιες ελιέ από τη Σεβίλη στην Ανταλουσία προς τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εδώ και 40 χρόνια έχουμε τέτοιες εξαγωγέ. Με επιχειρήσει πολύ σοβαρέ που δουλεύουν με μεγάλο επαγγελματισμό και που έχουν ε, ε, εδρεωθεί στις Ηνωμένε Πολιτείε και έχω επισκεφτεί και τα γραφεία του και τι εγκαταστάσει του εκεί. Γιατί λοιπόν αυτή η επίθεση τώρα ξαφνικά για μένα είναι φως φανάρι το πράγμα και αυτή η συμπάθεια που, και η συμπαράσταση που νιώθει ο κύριος Λουαζόν για το American First πάνω από όλα η Αμερική και αυτό το εθνικιστικό προστατευτισμό που επιβάλλουν αυτή είναι η κορυφή του παγόβονου. Θα, θα ακολουθήσουν και άλλα πολύ χειρότερα μετά. Γιατί μετά τις ελιές θα βρεθούν στο στόχαστρο και άλλες παραγωγές που ενδιαφέρουν περισσότερο τη Γαλλία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει που παράγονται τα προϊόντα αυτά, αν παράγονται στην Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, γιατί η κοινή γεωρική πολιτική είναι η ε, κοινή πραγματικά πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία και αφορά τις ενισχύσεις της ΚΑΠ και τις ενισχύσεις του greening. Έχουμε, το διακύβευμα είναι τεράστιο, δεν αφορά μόνο τις ελιές εδώ ή τις ισπανικές ελιές. Η νέα Αμερικανική κυβέρνηση επιβάλλει το νόμο της ε, και τους κανόνες της και όπου βλέπει παραγωγές ανταγωνιστικές θα, θα ε, ενεργήσει με τον τρόπο και το ύφος και το στυλ του κυρίου Τραμπ. Δεν, με αρκεί, δεν μου αρκεί η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περίμενα και περιμένω περισσότερα, ειδικά από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ξέρω ότι ενέχεται και η, Επιτροπή, και η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, αλλά και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Και χαίρομαι που ήρθε επιτέλους ο εκπρόσωπος περιμένω πολύ πιο πολεμοχαρή και μαχητική συμπεριφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντι στη ΣΥΠΑ. Γιατί μέχρι στιγμής παραίσασταν ευγενική ε, στη συμπεριφορά σας και διακριτική. Θέλω πιο μεγάλη μαχητικότητα και πυγμή. Και δεν ξέρω, ε, η Επίτροπος Μάλστρομ ή όποιος άλλος χρειαστεί ε, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το πρόβλημα. Γιατί αμφισβητούνται εδώ και δικηβεύονται οι εξαγωγές μας που την χάνουν ενισχύσεων με βάση την ΚΑΠ και που έχουν πάρει το πράσινο φως της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Και το χειρότερο είναι το ξέρουν αυτό οι Αμερικανοί. Γιατί πρόκειται για ένα σύστημα ουσιαστικά προστατευτισμού που θέλουν να εφαρμόσουν για τις παραγωγές τους, τίποτα παραπάνω. Και ελπίζω ότι ε, η, στην παρέμβαση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου θα αναφέρονται και κάποια επιπλέον μέτρα. Τι θα γίνει αν οι Αμερικανοί όπως αναμένεται, γιατί δεν τους ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα ούτε οι αναλύσεις. Όλα αυτά τα γράφω στα παλιά του στα παπούσια. Το, το μέτρο είναι πολιτικού χαρακτήρα. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα το υποστούμε. Ε, τότε περιμένουν σειρά και άλλες παραγωγές. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε καλύτερα τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και δεν μιλάω εδώ μόνο για τα ισπανικά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λοζό, ε, νομίζω ότι έχει διαφορετική πρόθεση με αυτά που είπε. Θα ξαναδώσω το λόγο στους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις δύο Γενικές Διευθύνσεις. Αποφασίστε μεταξύ σας Ποιο θα μιλήσει πρώτος και ποιος δεύτερος, αν θα μιλήσετε και οι δύο ή μόνο ένας, συνεννοηθείτε. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους βουλευτές για τα ερωτήματα που έθεσαν. Επιτρέψτε μου ε, να αναφερθώ λίγο στα όσα μόλις ε, είπε η κυρία Αγγιλέρα ε, Γκαρθία. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την ενίκηση άγκρη και εμπορίου. Έχουμε να κάνουμε με το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλε οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν συντονίσει τη θέση του. Και όπω σα είπα, ήδη έχουμε θετήσει μια συγκεκριμένη πολιτική στάση απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Και αντί απλώ να περιοριστούμε, όπω και σε πολλέ άλλε περιπτώσει, στο να παρέμβουμε ε, στην έρευνα ως ενδιαφερόμενο μέρος, ήδη έχουμε ε, δραστηριοποιηθεί σε πολιτικό επίπεδο απέναντι στη ΣΥΠΑ, ακριβώς μέσω γραπτών, γραπτής αλληλογραφίας και μέσω και άμεσης ε, προφορικής επικοινωνίας και μπορώ να σας πω πως το σύνολο των επιτρόπων, μάλιστα ειδικότερα προφανώς, έχει συζητήσει και έχει πάρει πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το ερώτημα του κυρίου ε, Λο, Ναι, ε, να να γίνει εδώ μια σκληρή, να δοθεί μια μάχη, αλλά αυτή θα δοθεί όταν θα έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά προ το παρόν κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην επιληθούν τα λόγω μέτρα. Και αυτό ακριβώ προσπαθούμε. Δηλαδή, εντό ε, του πλαισίου των κανόνων ε, ε, του ΠΟΕ προσπαθούμε, να, προσπαθούμε να πείσουμε την αμερικανική πλευρά ότι τα εν μέτρα δεν θα πρέπει να επιβληθούν. Τώρα, αν δεν τα καταφέρουμε να πείσουμε την αμερικανική πλευρά, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε κι εμεί. Ε, και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι πραγματικά είμαστε διατεθειμένοι να ε, δώσουμε εδώ μια σκληρή μάχη, όχι μόνο γιατί ε, θα βρεθούν σε δύσκολη θέση οι Ισπανοί παραγωγοί αλλά και επειδή θα προκύψει ένα συστημικού χαρακτήρα ζήτημα. Και εδώ, ποιο είναι αυτό το συστημικό ζήτημα, θα ήθελα να είμαι σαφής από αυτό. Δεν είναι ε, γεγονός ότι επειδή μια χώρα αποφασίζει να επιβάλλει κάποια μέτρα ε, κατά των ενισχύσεων ότι θα πρέπει εμείς ε, άμεσα να σταματήσουμε αυτές τις ενισχύσεις. Όχι, αυτό αποτελεί ένα μέτρο που λαμβάνει μια χώρα προκειμένου να αντισταθμίσει κατά την άποψή της, κατά εν λόγω ενισχύσεις. Και αυτό που είπε η συνάδελφος Γκονσάλες από την πλευρά δηλαδή ότι υπάρχουν, και συμφωνούμε εδώ ε, με τον ΠΟΕ, ότι υπάρχουν κάποια μέτρα ενισχύσεων τα οποία επιτρέπονται. Δεν έχουν στρεβλωτικό αντίκτυπο στην αγορά. Ενώ υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες ουσιαστικά καταστατηγούν τους ε, κανόνες έτσι ώστε να προσπαθήσουν να ε, ακυρώσουν τα όσα ισχύουν για τις ενισχύσεις από τη δική τους πλευρά όταν προέρχονται σε εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και όπως είπα αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει αυτή η έρευνα τη αμερικανική πλευρά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τα τεκτενόμενα, αλλά σας ε, διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή έχει ε, ενεργοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ. E, Σας ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, ήδη στείλατε επιστολές στην Επίτροπο Μάλμστρομ και στον Επίτροπο Χόγκαν. Οπότε έχουν ενημερωθεί αυτό το δύσκολο πρόβλημα και φαντάζομαι θα κάνουν τα απαραίτητα διαβήματα το συντομότερο δυνατό. Πάντως είναι πραγματικά χαρακτηριστικό το πώς ε, τα προστατευτικά μέτρα στο εμπόριο επηρεάζουν μονομένες χώρες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τώρα τους επισκέπτες ε, καλεσμένους του κυρίου Νίκολσον. Πρόκειται για νέους φοιτητές. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Και εμείς θα συνεχίσουμε στα δικά μας, στο επόμενο θέμα. Όπως θα καταλάβατε πριν από λίγο μιλήσαμε για τα προβλήματα που δημιουργούν οι πιθανές κυρώσεις των Αμερικανών εις βάρος των ε, Ισπανικών ελιών. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, την παρουσίαση της κατάστασης και των μέτρων για την καταπολέμηση ή τον έλεγχο της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων. Ένα ζήτημα που θίγει ιδιαίτερα τη Λιθουανία και την Πολωνία, αλλά και κάποιες γειτονικέ χώρες, αλλά και γενικώ στον κλάδο χείριου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να εξαπλωθεί αυτή η επιζώτια, γιατί κάτι τέτοιο θα επηρεάσει το εμπόριό μας και κυρίως το εξωτερικό μας εμπόριο. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό που αφορά την επιστημιστική ασφάλεια φυσικά, ένα ζήτημα ιδιαίτερα προσφυλές για τους καταναλωτές μας. Καλωσορίζω θερμότατα και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και θα δώσω πρώτα το λόγο στον Διευθυντή Bernard Van γνώριμο της ε, Επιτροπής μας. Θα σας δώσω το λόγο και από ό,τι ξέρω θα μας κάνετε μια παρουσίαση. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πόσα λεπτά έχω, 10 άντε 12. Θα προσπαθήσω να σας το πω σχετικά σύντομα, παρόλο που δεν είναι καθόλου απλό το θέμα. Θα... Έχουμε διάφορε διαστάσει στο φαινόμενο. Επιδημιολογική κατάσταση, περιφερειοποίηση που σύγχυε την Ευρωπαϊκή Ένωση, στρατηγική και κάποιε ευρωπαϊκέ δράσει. Καταρχήν, να δούμε την κατάσταση από το 2007 μέχρι το 2014. Θα δείτε παρακολουθώντας ε, το χάρτη ότι ξεκίνησαν τα κρούσματα από τη Γεωργία και το 2011, 2013 και 2014 εξαπλώθηκε η επιζωτία και σε άλλες χώρες. Βλέπετε γυρίζοντας πίσω πώς εξαπλώθηκε η ζωονόσος από τη Γεωργία αρχικά σε όλη τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και το 2014 έφτασε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμάστε ότι τα πρώτα κρούσματα ε, εντοπίστηκαν στα σύνορα με τη Λευκορωσία και υπάρχουν πια κρούσματα στην Πολωνία, Λιθουανία, Λετωνία και Εστονία. Οι πράσινες κοιλίδες στην οθόνη δείχνουν τα κρούσματα σε κτηνοτροφικές μονάδες και τα κίτρινα, ε, οι κίτρινες κοιλίδες ε, αφορούν αγριογούρουνα, αγριογούρουνα που βρέθηκαν νεκρά και τα κουφάρια τους διαγνώστηκαν με αφρικανική πανόλη των χείρων. Ε, βλέπετε και άλλους χάρτες με την εξάπλωση της ζωονόσου που πέρασε από τα σύνορα και επεκτάθηκε και στην ενδοχώρα των Βαλτικών χωρών και της Πολωνίας. Η κατάσταση στην Ευρώπη τώρα βλέπετε την επισκόπηση από τα έτη 2016 και 2017. Έχουμε πολλές πράσινες κοιλίδες, αλλά και κυτρινές μεταγριογούρουνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα εξέτασης και των αγριογούρων που δεν ε, υπάρχει αντίστοιχο στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές πράσινες κοιλίδες. Δεν σημαίνει ότι μόνο εμείς έχουμε πράσινες κοιλίδες, αλλά επειδή μόνο εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα, εντοπίζουμε τα κρούσματα και στα αγριογούρουνα. Να... Θα μιλήσω αργότερα για τις τέσσερις πληγήσεις χώρες μέλη να σας κάνω μια μικρή παρουσίαση πέραν το τι συμβαίνει στην Τσεχία και που συνέβη το καλοκαίρι που πολύ κοντά στο δρόμο βρέθηκε ε, μολυσμένο αγριογούρουνο. Φαίνεται λοιπόν ότι η εξάπλωση έγινε από ανθρώπινο παράγοντα, ίσως από κάποιο τελικέρι που μετέφερε σαλάμι ζαμπόν από την Ουκρανία και το άφησε στο πάρκινγκ, στη στάθμευση που ε, έμεινε το βράδυ. Είχαμε εξάπλωση της επιζώτιας. Ο ανθρώπινος παράγων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στοιχείο της μετάδοσης. Βλέπετε εδώ το χάρτη με μία μόνο κοιλίδα στη Τσεχία, γιατί 50 αγριογούρουνα εντοπίστηκαν σε πολύ μικρή περιοχή που τη βλέπετε στο χάρτη. Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα, ειδικά στη Τσεχία, είναι η συμπεριφορά των κυνηγών. Οι κυνηγοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν πραγματικά στην εξάλληψη της ε, ζωονόσου. Ή το αντίθετο θα μπορούσαν να συμβάνουν στην εξάπλωση της επιζώτιας σε πολύ ευρύτερες περιοχές. Στη Τσεχία Πάντως έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις οργανώσεις κυνηγών και μέχρι στιγμής καταφέραμε να περιορίσουμε την ζωονόσο μόνο στα αγριογούρουνα και μάλιστα σε μια πολύ μικρή περιοχή. Βλέπετε από τον Ιούλιο τον αριθμό των κρουσμάτων ανά εβδομάδα. Άκρα δεξιά έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις μολυσμένων αγριογουρούνων ελπίζουμε με συνέχιση των προσπαθειών στην Τσεχία να εξαλείψουμε πλήρως την επιζώτια αυτή. Περνάμε στη Ρουμανία. Εκεί είχαμε δύο περιπτώσεις στη Ρουμανία, σε δύο βλές που βρέθηκαν αμολισμένα ε, γουρούνια, αλλά όχι αγριογούρουνα και πάλι ανθρώπινο παράγοντα από παράνομη εισαγωγή ε, κρέατος και μεταποιημένων υπολοιμάτων φαγητών που δόθηκαν σε χείρους. Ε, βέβαια, χάρη στην καλή συνεργασία με τις ρουμανικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, δεν είχαμε εξάπλωση τη ζωονόσου πέραν αυτών των δύο περιπτώσεων, που σε δύο αυλές, ε, σε πολύ μικρές περιπτώσεις είχαμε αυτά τα κρούσματα. Οπότε θεωρείται λήξαν το ζήτημα της Ρουμανίας. Και πάλι εδώ έχουμε τη χαρτογράφηση για τη Ρουμανία και σε ένα χάρτη βλέπετε ότι είναι σε ένα προάστιο ουσιαστικά και επειδή ήταν ακριβώς περιορισμένη η περιοχή, διευκολύθηκε το έργο των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Τώρα βλέπουμε τα κρούσματα από την αρχή του 2017. Στη Τσεχία είχαμε πολλά αγριογούρουνα, αλλά επαναλαμβάνω σε πολύ περιορισμένη περιοχή γεωγραφική, σε ένα δάσο ουσιαστικά, μικρό, ενώ τα υπόλοιπα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Πολωνία και στις τρεις χώρες της Βαλτικής. Στη Ρουμανία είχαμε μόνο δύο περιπτώσεις χείρων, κόσιτων. Τώρα, τι ε, μέτρα αναλάβαμε από την αρχή ε, της επιζωτίας. Και εδώ πάλι σύντομα να δούμε κάποιους χάρτες από τα μέσα του 2014 όπου είχαμε τα πρώτα κρούσματα σε αγριογούρουνα από τη Λευκορωσία που μόλυναν ζώα και στην Πολωνία και η Λιθουανία. Μετά υιοθετήσαμε την αρχή της περιφερειοποίησης που έγινε δεκτή από κάποιες τρίτες χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά αλλά όχι και από άλλες χώρες όπως η Ρωσία που από εκεί έχουμε απαγόρευση από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για χείριο κρέα. Έχουμε τελείω διαφορετική δηλαδή κατάσταση και αντίδραση των εταίρων μα. Εδώ βλέπουμε την εξέλιξη της ζωονόσου από το 2014 μέχρι σήμερα. Τα μπλε τμήματα είναι ε, αυτές οι ζώνες προστασίας ε, ε, που έχουμε κάποιες, κάποια κρούσματα, αλλά όχι αγριογούρουνα. Στα, στις ροζ περιοχές έχουν μολυθεί και αγριογούρουνα και στις κόκκινες περιοχές έχουμε σε εκμεταλλεύσεις μόνο. κόκκινα λοιπόν εκμεταλλεύσεις, ροζ αγριογούρουνα και Buffer zone είναι το γαλάζιο. Προφυλακτήρα, αν θέλετε, προσπαθούμε να αρχιετήσουμε την επέλαση και στις υπόλοιπες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπετε την εξέλιξη από το 2014 και μετά. Τώρα, αν αποκλείσουμε τα πιο σημαντικά, που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως σας ανέφερα, αν εφαρμόσουμε στην επιζωτία πιστά τις συστάσεις ε, για τη διαχείριση της άγριας πανίδας. Η εξάπλωση της νόσου θα είναι ένα χιλιόμετρο το μήνα. Δυστυχώς όμως, σε μερικές περιοχές, η συμπεριφορά των κυνηγών ε, δυστυχώς δεν ήταν συμβατή με τις συστάσεις και όπως είδατε και από την εξέλιξη στους χάρτες είχαμε δυστυχώς δραματική εξάπλωση της ζωνός τα τελευταία χρόνια. Οπότε ανακεφαλαίωση. 36 ε, εφαρμοστικές αποφάσεις. Ε, ήρθε η ώρα για αναθεώρηση της κατάστασης με τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων. Ποια είναι η στρατηγική μας. Δύο κυρίως σκέλη. Διαχείριση των, για, και εδώ κέρια σημασία έχει συμπεριφορά των κυνηγών για να αποφευθεί η εξάπλωση της σου και ανθρώπινος παράγων. Πρόκειται για ανθρώπους που χωρίς να το γνωρίζουν ή χωρίς να έχουν συνείδηση θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εισαγωγή κρέατος ή κάνοντας προσωπικές ε, ε, προσωπικά εισαγωγές ε, προϊόντων από περιοχές που έχουν μολυνθεί από την όσο. Και το λέω γιατί ε, με εξαίρεση την Τσεχία και τη Ρουμανία όλα τα κράτη-μέλη που δεν είχαν αναμειχθεί μέχρι στιγμής έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, έχουν λάβει τις προειδοποίησεις για να επισημάνουν το πρόβλημα στους κυνηγούς, στους δελικέριδες, στους δασοκόμους, ακόμη και σε εργαζομένους σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Θέλουμε να γίνει μια ενημέρωση και στις χώρες που δεν έχουν πληγή για να συνειδητοποιήσουν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι ότι όταν εισάγουν προϊόντα, ακόμη και σαλάμι ζαμπών, ακόμη ε, και στα παπούσια τους μπορεί μερικές φορές να εντοπιστεί και να παραμείνει ο ιός που είναι πολύ ανθεκτικός. Θα πρέπει να γίνει μια γενική συνειδητοποίηση και στις χώρες που ακόμη δεν έχουν μολυνθεί. Τώρα, στα πλαίσια της α, ε, οργάνωσης που λέγεται GFTDS, οργανώσαμε συντονιστικές συνεδριάσεις για να θετήσουμε μια συνεκτική στάση με τις ε, εμπλεκόμενες χώρες, όχι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά και τη Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία και Μολδαβία. Και όπως βλέπετε αφιέρωσαμε διήμερε συνεδριάσεις ε, για σημαντικά θέματα όπως είναι η διαχείριση των ε, αγρογούρων, των οικόσιτων χείρων και ε, τους τελευταίους μήνες ασχοληθήκαμε με το θέμα της ε, επικοινωνίας και της ε, συνειδητοποίησης που θα πρέπει να λάβει η χώρα της ενημέρωσης. Εφτά ήταν οι θυγήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, τρεις της Βαλτικής, Ουκρανία, Πολωνία, Λευκορωσία και Ρωσία και κάναμε επισκέψεις και στις υπόλοιπες χώρες για να γίνει ενημέρωση και γνώση της κατάστασης. Επίσης έχουμε εμπειρογνώμονες και για, την, για τα αγριογούρουνα και για, τα, 20, τα τους με επισκέψεις ώστε να ενημερωθούν οι ενεχόμενες χώρες και η Τσεχία και η Ρουμανία όταν είχαμε τα κρούσματα και σε αυτές τις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ορμόδιος Επίτροπος Ανδριοκάητες ε, οργάνωσαν τέσσερις ε, υπουργικές συναντήσεις υψηλού επίπεδου, ήδη έχουν γίνει τέσσερις. Η επόμενη θα γίνει στην Πράγα σε κανένα δύο μήνες και επίσης σε υπουργικό επίπεδο είχαμε 10 υπουργούς που παρέστησαν στις συνεδριάσεις αυτές και πάλι για να ε, γίνει ενημέρωση και συνειδητοποίηση του προβλήματος και να ενημερωθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για να παρακολουθήσουν τις και να ακολουθήσουν μάλλον τις κατευθυντήριες γραμμές. Τώρα, Παγκόσμιο Οργάνωση Εμπορίου, ε, Επιτροπή Προσφυγών. Κατά την καταγραφή των πρώτων κρουσμάτων στις χώρες Βαλτικής και την Πολωνία, η Ρωσία αποφάσισε να απαγορεύσει τις αγωγές χείριου κράτους από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλος χερός. Κάτι που δεν είναι αποδεκτό από εμά φυσικά. Γι' αυτό και καταθέσαμε αγωγή στην Επιτροπή Προσφυγών στη Γενέβη και μάλιστα κερδίσαμε το πρώτο τμήμα. Η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου ε, αναγνώρισε ότι θα, η περιφερειοποίηση που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αρκεί για να προστατεύσει το εμπόριο. Οπότε η Ρωσία είναι υποχρεωμένη να άρει την απαγόρευση εισαγωγό χείριου κρέατος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα 6 ε, Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία. Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να ξανανοίξει τις αγωγές χείριου από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν το κάνει θα συνεχίσουμε την προσφυγή μας στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου με βάση τις κανονικές διαδικασίες. Τώρα, ε, παρέχουμε υποστήριξη όχι μόνο α, ε, στις, ε, στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις γειτονικές χώρες μέσω workshop ε, και από εκεί και μετά μέσω τεχνικών αποστολών υποστήριξης και εδώ αναφέρομαι ε, ειδικότερα στο, στην κτηνιατρική ομάδα έκτακτης βοήθειας, ε, ειδικότερα εδώ αναφέρομαι ε, σε μια ομάδα η οποία αποτελείται από 21 εμπειρογνώμονε, οι οποίοι επιτόπου πιστεύουν τα κράτη-μέλη για να δώσουν συμβουλέ ω προ το πώ θα πρέπει να αντιδράσουν και τι θα πρέπει να κάνουν, όπω για παράδειγμα όταν υπήρξε ένα κρούσμα στη Ρουμανία. Από εκεί και μετά υπάρχει και παροχή συμβουλών από την ΕΦΣΑ, την αρχή δηλαδή για την ασφάλεια των ε, τροφίμων. Υπάρχει και το εργαστήριο αναφοράς ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει αντιδραστήρα στα, στις χώρε. χώρες. Από εκεί και μετά έχουμε οικονομική υποστήριξη που παρέχεται για την εξαγωγή προγραμμάτων, όχι μόνο στα κράτη-μέλη εκείνα όπου υπήρξαν κρούσματα της ασθένειας, αλλά και σε όλα τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν σύνορα με αυτά τα κράτη-μέλη, δηλαδή από τη Φιλανδία ως τη Ρουμανία. Επίσης υπάρχουν και κάποιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινή γνώμης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αγριόχειρων, την αποζημίωση των ε, γεωργών, ε, στα κράτη-μέλη τα οποία πλήγησαν από κρούσματα. Και εδώ βλέπετε και ένα πίνακα ε, με τα συνολικά ποσά συγχρηματοδότησης θα διαπιστώσετε ότι από το 2013 υπάρχει αυτή η συγχρηματοδότηση, δηλαδή ήδη πριν από το πρώτο κρούσμα το οποίο σημειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε υποστήριξη υποστήριξη ε, προς τα κράτη-μέλη που είχαν, ε, βρίσκονταν στο μεγαλύτερο κίνδυνο. Και το σύνολο αυτή τη χρηματοδότηση που έχει διατεθεί μέχρι στιγμή φτάνει τα 36 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και μετά υπήρξε ε, συγχρηματοδότηση και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βέβαια ο στόχο μα είναι να μην εισέρχεται καν αυτή η ασθένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε χρειάστηκε να γίνουν κάποιε δαπάνε σε χώρε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκίνησε λοιπόν κάποιας, ε, κάποια πιλωτικά προγράμματα που έχουν ξεκινήσει στην Μολδαβία και την Ουκρανία. Ε, από εκεί και μετά υπάρχουν ε, μια σειρά από έλεγχοι που λαμβάνουν χώρα από τους δικούς μας ελεγκτές. Ο τελευταίος πριν από το καλοκαίρι έλαβε χώρα από την πλευρά των ελεγκτών μας σε όλες τις χώρες της στα ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου ακριβώς να υπάρξει περισσότερη ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά τους κατάλληλους συνοριακούς ελέγχους ε, και στη Φιλανδία ή μάλλον από τη Φιλανδία ως τη Ρουμανία, ώστε να διασφαλίζεται ότι όσοι ε, επιστρέφουν από τα ταξίδια τους ε, που κάνουν στη Ρωσία, στη Λευκορωσία, στη Μολδανία και την Ουκρανία έχουν ενημερωθεί αρκούντως σε ό,τι αφορά τους κινδύνους της μεταφοράς ε, κρέατος από αυτές τις χώρες. Γιατί είδατε βέβαια ότι σε εκείνες τις χώρες σημειώθηκαν πολλά από τα κρούσματα. Εάν μου επιτρέπετε ένα ακόμα λεπτό θα κάνω μία σύντομη ε, σύνοψη εδώ, τρεις διαφάνειες ακόμα μου έχουν ε, ε μείνει. Ε, η λάμπη skin disease, η οποία έχει σημειωθεί δηλαδή με κάποια κρούσματα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και έχει αρχίσει να, από το 2016 να εξαπλώνεται και ε, υπάρχει βέβαια ήδη και ένα εμπόλιο κατά του λαμπισκίν ε, το οποίο ήδη έχει αναπτυχθεί και είναι πολύ αποτελεσματικό και έτσι λοιπόν εμείς έχουμε παράσει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμβόλια σε όλες τις χώρες που είναι σε μπλε χρώμα δηλαδή ε, Σκόπια, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σερβία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση. και μάλιστα υπήρξε ε, και μια υπουργική διάσκεψη με τον ε, Επίτροπο Αντριουκάτη, στην οποία παρευρέθηκαν 15 υπουργοί από την Ιταλία στην Αυστρία και ε, καλύπτοντα όλο το, τα Βαλκάνια και το νότο εδώ τη Ευρώπη. Με αυτέ λοιπόν τι κοινέ προσπάθειε καταφέραμε να σταματήσει εκεί που βρισκόταν η ασθένεια και έχουμε δυόμιση ε, εκατομμύρια δόσεις εμβολίων ε, ως ε, απόθυμα που έχουμε δημιουργήσει και τα οποία μπορούν να αποστολούν σε όλες αυτές τις χώρες των Βαλκανίων και φυσικά και στην Ελλάδα. Και όλες αυτές λοιπόν οι προσπάθειες μας οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ, δηλαδή νωρίτερα φέτος, όπου είναι η Αλβανία η μόνη χώρα όπου σημειώνονται κρούσματα. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες δεν υπάρχουν κρούσματα μέσα στο 2017 της οριζόντου δερματίτης του Λαμπισκίν, ε, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ακριβώς ότι ο συντονισμός στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κίνητρα τα οποία δόθηκαν στα κράτη-μέλη μέσω ακριβώ ε, και αυτή τη ε, τοποθέματο εμβολίων οδήγησαν τελικά στην αποτροπή τη περαιτέρω εξάπλωση τη ασθένεια σε άλλε χώρε όπω η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Κροατία και άλλοι. Ε, τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τη βλέπετε εδώ στο χάρτη, με βάση την οποία ε, μάλλον κυκλοφορεί ο ιός ακόμα και ε, σε κίτρινο βλέπετε τις περιοχές εκείνες όπου δεν έχει εντυπιστεί ο ιός. Ε, και τώρα με τις 15 ε, δεθυγόμενες χώρες θα γίνει μια κοινή ε, συνεννόηση ούτως ώστε να αποφασίσουμε την στρατηγική μας για το επόμενο έτος η οποία θα περιλαμβάνει πιθανότητα ένα νέο εξολοκλήρωμένο εμβολιασμό προκειμένου να διασφαλίσουμε την πλήρη εξάλληψη της ασθένειας από το 2019 και μετά. Αυτά λοιπόν εν ολίγης ως προς τα όσα έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά το Λαμπίσκιν. Αυτά ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε στην αίθουσα και εκπροσώπους της α, Κλαδικής Ομοσπονδίας από την Πολωνία και τον αντιπρόεδρο της Κοπακοζέκα. Κύριε Σράιερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στις ε, κάτω χώρες ε, το 1997, έζησα από κοντά αυτή την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Ήταν τραγική η κατάσταση. Θα πρέπει να συγκρατηθεί η επιδημία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ε, πρέπει να πω όμως ότι και την προηγούμενη φορά που είχαμε μια αντίστοιχη συζήτηση ακούσαμε πολλές ε, ε, συζητήσεις και άκουσα και πολλές επικριτικές τοποθετήσεις εναντίον των κυνηγών. Υπήρχαν μερικοί μάλιστα που έλεγαν ότι θα πρέπει το κυνήγι να απαγορευτεί γιατί είναι τα αποτέλεσμα τα αρνητικά. Εδώ τώρα όμως ακούω από εσά ότι μπορεί να παίξουν και θετικό ρόλο οι κυνηγοί. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Γίνεται λόγος ε, για την Πολωνία και αν ε, ε, γνωρίζω καλά την κατάσταση καταλαβαίνω ότι κινούνται πολύ, μετακινούνται πολύ σε όλη την Ευρώπη οι κυνηγοί. Άλλη ερώτηση. Η προσέγγιση όσον αφορά την ασθένεια αυτή, την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων δηλαδή, είναι εναρμονισμένη η προσέγγιση, γιατί παλιά δεν ήταν. Ε, επίσης, εισαγωγές ε, χειρίου κρέατος ε, στην Ρωσία. Συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε το θέμα. Όσον αφορά τώρα τα αγριογούρουνα ε, από ό,τι φαίνεται στην ε, Ρωσία ε, έχουν σκοτώσει όλα τα αγριογούρουνα. Αυτό είναι η κατεξοχήν ας πούμε προληπτική δράση και μέτρο. Η άποψή σας εσάς ποια είναι όσον αφορά το θέμα αυτό. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν ξέρω και πολλά πράγματα για αυτά, δεν έχουμε πολλά αγριοπούρουνα. Ε, Έχουμε μερικά τα οποία έχουν ξεφύγει από τις ε, ε, φάρμες, από τις ε, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Φαίνεται πάντως ότι πρόκειται εδώ για μια ασθένεια η οποία είναι και σοβαρή και εξαπλώνεται πολύ. Θα ήθελα όμως να πω μήπως και το θέμα με τα κουνέλια που έχει προκύψει ε, ίσως ε, μας έχει διδάξει ότι αυτές οι επιζωτίες ε, έχουν μια κυκλική ας πούμε ζωή. Επίσης, αυτό μας έμαθε τουλάχιστον η μιξομάτωση των κουνελιών. Ε, φαίνεται πάντως ότι στην προκείμενη περίπτωση της Αφρικανικής Πανόλης ε, δεν υπάρχουν ε, σημαντικές δευτερογενείς επιζώτιες. Επίσης, να ρωτήσω το εξής. Στις βαλτικές χώρες και στην Πολωνία οι αρχές κοινοποιούν το γεγονός ότι ε, οι Πολωνοί εργαζόμενοι που πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να μεταδώσουν την ασθένεια αυτή και λαμβάνονται μέτρα για να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Ε, επίσης ε, γίνεται εσείς βέβαια είστε πληρωμέ, πληρώνεστε για να αναφερθείτε και σε ενδεχόμενη θεραπεία της οζόδους δερματίτιδας. Υπάρχει κανονική θεραπεία, υπάρχει εμβόλιο θα προσπαθήσετε να προσπαθήσετε επίσης να σκοτώσετε όλα τα αγριογούρουνα ε, στις, ε, ε, στα σύνορα, στις μεθοριακές, διασυνοριακές έτσι, περιφέρειες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ που συμπεριλάβατε και αυτό το θέμα στην ημέρη σε διάταξη και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πλήρη ενημέρωση που μας έκανε ως προς το θέμα αυτό. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω κάτι τέτοια. Τρίτη φορά είναι που εγκύπτουμε στο θέμα αυτό και επιτέλους φαίνεται να εξετάζει κάποια μέτρα για να εξαλείψει την επιζωτία, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι και πολύ θετικά. Από το 2014 και μετά είχαμε μια επιδείνωση της κατάστασης και οι της χώρας δεν έχουν βρει κάποια αποτελεσματικά μέτρα για την εκρίζωση της ασθένειας. Εκεί είχαμε στη Λιθουανία το 2014 κάποια κρούσματα, ενώ σήμερα τα δύο τρίτα ε, του, της επικράτειάς μας έχει παρουσιάσει κρούσματα εκτεταμένα τέτοιας επιζώτιες. Και μάλιστα οι μικρές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αδυνατούν πια να ασχοληθούν με χειροτροφία. Οπότε ε, δεν έχουμε και αυτάρκεια. Το 50% του χείριου το εισάγουμε. Οπότε αν δεν έχουμε δυνατότητα ούτε καν να εισάγουμε θα παρουσιαστεί έλλειψη χειρίου κρέατος στη Λιθουανία. Προτάθηκε αντικατάσταση του χείριου κρέατος από το βόιο. Βέβαια, βάσει κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούμε να αυξήσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο ε, βοηδών, ούτε καν το ζωικό κεφάλαιο προβάτων, γιατί κάτι τέτοιο αντιβαίνει στους ε, ισχύοντες κανόνες. Οπότε, ναι, με δεν μπορούμε να ε, εκθρέψουμε χείρους, αλλά δεν μπορούμε να αυξήσουμε ούτε το ζωικό κεφάλαιο ε, βοηδών και προβάτων. Βρισκόμαστε σε διέξοδο λοιπόν, γιατί μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε κρέας. Επίσης παραλείψατε κάποια σημαντικά ε, γεγονότα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2014 εντοπίστηκε μια μεγάλη αιστεία της ζωνόσου στη Λιθουανία. 20%, 20.000 μάλλον ε, χείροι χρειάστηκε να θανατωθούν και πριν από λίγους μήνες είχαμε πάλι θανάτωση 24.000 χείρων. Ε, θανάτωση και ταφή. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί όμως ότι τα μέτρα αυτά είναι αποτελεσματικά και θα αρκέσουν για την εξάλληψη της ε, ζωονόσου, ακόμη και στις ε, ε, εντατικές κτηνοτροφικές μονάδες. Στις μικρές ούτε συζήτηση. Επίσης, ε, δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα αίτια της μόλυσης, ποιες είναι οι πηγές ε, της μόλυσης. Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται αυτή η νόσος. Λέτε ότι μπορεί να μεταδοθεί και από σαλάμι, από ζαμπόν. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα τώρα. Νομίζω ότι διαπιστώνουμε αναποτελεσματικότητα των μέτρων, διαπιστώνουμε επιδίνωση της κατάστασης, αλλά μένουμε ανήμποροι. Σε λίγα χρόνια ολόκληρη η Πολωνία θα έχει μολυνθεί από την, ε, πανόλη, την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Θα πρέπει να περιμένουμε να εξαπλωθεί ε, η ζωονόσος και στη, μέχρι τη Γαλλία και τη Γερμανία για να αναλάβουμε επιτέλου αποτελεσματικά μέτρα. Και από τη στιγμή που σήμερα οι αγριόχειροι θεωρούνται ε, φορείς, γιατί θα πρέπει να αφήνουμε τη λύση μόνο στα χέρια των κυνηγών. Είναι γελίο. Οι κυνηγοί ενδιαφέρονται για πολλά ζώα. Δεν θέλουν να εξολοθρεύουν ή να θανατώνουν συγκεκριμένο είδος. Ούτε τους ενδιαφέρουν τα θηλυκά καταρχήν ζώα τους κυνηγούς, μόνο στα αρσενικά στοχεύουν. Οπότε ξοδέψατε πόσα, 5 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά, 10 εκατομμύρια τη δεύτερη. Το 2017 θα χρειαστούν 36 εκατομμύρια και σε 5-10 χρόνια θα χρειαστούν ακόμη υψηλότερα κονδύλια για να αναχαιτήσουμε την εξάπλωση της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων. Επίσης, μας είπατε ότι στη Τσεχία και τη Ρουμανία η ζωονόσος αυτή έχει σχεδόν εξαλειφθεί δεν σας πιστεύω. Γιατί στη Λιθανία ακούσαμε πολλά λόγια, έγιναν εκτεταμένες συζητήσεις, αλλά αποτελέσματα δεν βλέπω. Θα πρέπει επιτέλους να επιβάλλουμε υποχρεωτικά κάποια μέτρα και να συμφωνήσουμε και να εφαρμόσουμε έναν οδικό χάρτη. Γιατί αν αδρανίσουμε σήμερα, η κατάσταση στο μέλλον θα είναι πολύ χειρότερη. Ο συνάδελφος είπε ότι η νόσος αυτή, η νόσος, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ισχύει όμως αυτό. Αυτή η πληροφορία είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Θέλω να βρούμε αποτελεσματικά μέτρα και μηχανισμούς για να μας επιτρέψουν να εξαλείψουμε την νόσο αυτή. Ο κύριος Μπούντα. Παρακαλώ μην μυθείτε τον προλαλήσαντα και τηρήστε το χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία και στην Ρουμανία είχαμε επίσης τέτοιες εστίες. Εγώ θέλω συγκεκριμένα να μου πείτε πώς είναι δυνατόν να σταματήσουμε την μετακίνηση των αγρίων ζώων. Μα τα αγρία ζώα δεν ξέρουν από σύνορα για να σταματήσουν εκεί. Ε, υπάρχουν ε, προβλήματα με τα ε, άγρια ζώα τα οποία περνούν τα ε, σύνορα. Έχετε σκεφτεί ας πούμε να βάλετε στα σύνορα εκεί που ξέρετε ότι τα, οι αγριόχειροι χρησιμοποιούν κάποια σημεία ως πέρασμα στα περάσματα αυτά να βάλετε ενδεχομένως κάποια ηλεκτροφόρα σύρματα. δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εμπιστευόμαστε και τόσο τυφλά ε, τους ε, ε, κυνηγούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ληφθούν άλλα μέτρα. Βεβαίως για το προσωπικό του συμφέρον οι κυνηγοί θέλουν να σκοτώσουν όσο γίνεται περισσότερα αγριογούρουνα αλλά ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουμε ε, κάποια κατόφλια έτσι ώστε να μην φτάσει η αρρώστια μέχρι τη Γερμανία. Κύριε Πετήρ, ευχαριστώ. Εμείς ευτυχώς στην Κροατία δεν έχουμε τέτοια κρούσματα. Και μάλιστα είχαμε πρόβλημα με την αύξηση του πληθυσμού των αγριόχειρων που πολλαπλασιάστηκαν τόσο πολύ σε μερικές περιοχές που φτάνουν στις αυλές, καταστρέφουν τις καλλιέργειες και οι γεωργοί μας δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τέτοια εξάπλωση αγριόχειρων. Εμείς έχουμε κάποιες αρχές οικονομικές αλλά δεν ε, έχουμε ξεχωριστό αριθμό για, τα, για τους αγριόχειρους που μερικές φορές διασταυρώθηκαν με ήμερα γουρούνια και αυξήθηκε ο πληθυσμός τους. Πάντως, τι μέτρα μπορούν να λάβουν χώρες που δεν έχουν ακόμη πληγή και πώς μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των, αγρι, των αγριόχειρων ώστε να επιτρέψουν στους γεωργούς τους να προστατεύσουν τις καλλιέργειες και τις πορές τους. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Και θα ήθελα να υποβάλω και εγώ μια ερώτηση. Επι, επιμελητιακά, πώς αντιμετωπίζετε το θέμα. Ε, θα, έχουν καταρχήν να θανατωθεί μεγάλα κοπάδια, γιατί ο κλάδος είναι ιδιωτικοποιημένος. Ε, δεν ξέρω τι προθυμία έδειξαν οι κτηνοτρόφοι για θανάτωση πως επιμελητιακά εφαρμόστηκαν τα μέτρα. Επίσης, πώς θα αποτρέψουμε την περαιτέρω εξάπλωση αυτής της νόσου. Επίσης, ε, η νόσος αυτή έπληξε κυρίως μικρές ε, εκμεταλλεύσεις που δεν είναι σε θέση να τηρήσουν τις ε, προϋποθέσεις είναι απροετοίμαστες ε, οι μικρές κτηνοτροφικές μονάδες ε, για να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα της ασφάλειας και να αποτρέψουν την εξάπλωση της ζωνόσου. Και μάλιστα ε, οι χώρες αυτές που είναι κυρίως νέες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ ανεπτυγμένη χειροτροφία μικρής κλίμακος και γι' αυτό ήταν δύσκολη η αντιμετώπιση από τους μικρούς, ε, μικρής κλίμακας αυτής κτηνοτρόφους αντιμετώπιση του προβλήματος. Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση. Αν κάποιος θανατώσει, για παράδειγμα, ένα μικρό κοπάδι χείρων που έχει, έχει δυνατότητα να λάβει ενίσχυση επενδύσεις ε, σε άλλα ζώα κρεατοπαραγωγής. Φαντάζομαι ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης ε, για έναρξη νέας ε, μορφής κρεατοπαραγωγής σε περίπτωση θανάτωσης του κοπαδιού σε τέτοιες μικρές κτηνοτροφικές μονάδες. Γιατί έχει διατυπωθεί ανησυχία και φόβος ότι θα εξαπλωθεί περαιτέρω αυτή η επιζώτια τι μέτρα επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί και να αναχαιτιστεί αυτή η νόσος. Ευχαριστώ και θα σας δώσω και πάλι το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να σας πω Δύο λόγια πρώτα απ' όλα για τα αγριγούρουνα. Όπως είπατε και προηγουμένως, ε, η προετοιμασία και η πρόληψη είναι απολύτως ε, σημαντικές έτσι ώστε να αποφευχθεί η ε, διάχυση της ασθενείας. Αυτό είναι σημαντικό για όλους. Θα πρέπει να κατανοήσουν και οι κτηνοτρόφοι πώς ε, μπορούν να αυξήσουν την βιοασφάλεια ε, ε, της φάρμας τους. Αυτή η, η διάχυση, αυτό το spider effect μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το ξέρουν. Και δυστυχώς όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι μεγάλες κτηνοτροφικές ε, μονάδες, υπήρξαν μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες αναγκάστηκαν να θανατώσουν ε, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ε, χείρων. Όσον αφορά την παρατήρηση του κ. Άγνιου, γνωρίζω ότι δεν υπάρχουν αγριογούρουνα Καλά, καλό είναι αυτό και για την ε, ε, Μεγάλη Βρετανία και για τη Δανία όπου βλέπουν τα χρεογρούνα μόνο στους ζωολογικούς κήπους. αλλά και στις χώρες αυτές ε, θα πρέπει να επαγρυπνούν οι κτηνοτρόφοι και εν πάση περιπτώσει οι εργαζόμενοι της κτηνοτροφίας, οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή χρησιμοποιούν ζαμπόν ή σαλάμι θα πρέπει να ε, ε, είναι ενημερωμένοι, αλλά και αυτοί που περπατούν στα δάση. Ε, μπορεί να κουβαλήσουν λάσπη ε, στις ε, μπότες τους, στα παπούτσια τους και πολύ συχνά αυτοί οι οποίοι πάνε να μαζέψουν μανιτάρια, δραστηριότητα πάρα πολύ διαδεδομένη, μπορεί να προκαλέσουν την μετάδοση του ιού. Εν πάση περιπτώσει για να προληφθεί ή να αποφευθεί η διάθεση πρέπει να αποφευθει η διαθεση πρεπει να αντιμετωπισουν και το ζήτημα των αγριοχείρων ε, και ε, έτσι ώστε να αποφευχθεί ε, μεγάλο οικοφορτίο φορτίο στα δάση. Έχει αποδειχθεί σε, ε, χώρες, ε, σε πολλές χώρες ε, ότι όταν μειώνεται αυτό το οικοφορτίο φορτίο και όταν δηλαδή κανείς απομακρύνει τα κουφάρια των αγριογούρων έγκαιρα από τα δάση τότε μειώνεται η πιθανότητα μετάδοσης. Όσον αφορά το εμβόλιο, ναι πράγματι δεν υπάρχει εμβόλιο. Είμαστε πολύ κοντά βέβαια δεν το ανέφερα προηγουμένως στην παρουσίασή μου, εκατομμύρια δαπανούμε ε, στην έρευνα έτσι ώστε να βρεθεί ε, αυτό το ε, εμβόλιο αλλά εν πάση περιπτώσει στο εγγύς μέλλον δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Είναι γεγονό πάντως ότι η ασθένεια αυτή δεν παρουσιάζει επιπλοκές ή οποιαδήποτε, δεν έχει οποιαδήποτε ε, συνέπεια στην ε, ανθρώπινη υγεία και δεν είναι πολύ επικίνδυνη. Ρουμανία τώρα, δυστυχώς έφυγε ο Ρουμανός βουλευτής, αλλά φαίνεται ότι πέρασε ε, η ασθένεια αυτή και έληξε ε, ε, στις ημιαστικές, περιαστικές μάλλον περιοχές είχαμε κάποια κρούσματα, τώρα δεν υπάρχουν πια. Όσον αφορά την Ρωσία, εγώ θα αναφερθώ στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Στην Λευκορωσία δεν έχουν αγριοχείρους. Έτσι μας είπαν, αλλά δύσκολα το πιστεύουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά ε, τους ε, πείσαμε να παραδεχτούν ότι έχουν και αγριόχειρους. Και εμεί ξέρουμε, αλλά είπανε δεν έχουν ε, κρούσματα της ασθένειας, αλλά εμεί ξέρουμε ότι έχουν κρούσματα. Και τους είπαμε ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν. Πολλές χώρες έχουν, αυξηθεί, έχουν αυξήσει συγγνώμη, την, το κυνήγι των αγρίων χείρων. και φέτος ε, είχαμε περισσότερη, περισσότερο κυνήγι ε, από άλλες χώρες. Αυτό μπορεί πράγματι να βοηθήσει. Όσον αφορά τη Γενέβη, το είπα και προηγουμένως, ε, οι Ρώσοι έχουν ε, προθεσμία να συμμορφωθούν μέχρι την 6η Δεκεμβρίου και αν όχι εμείς θα προχωρήσουμε με τις προσφυγές ενώπιον του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου που κάθεται δίπλα μου, έτσι ώστε να προσπαθήσει να σας εξηγήσει ποια, ε, εν συντομία ποια είναι η στρατηγική μας για τους ε, γιατί αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι και ο ρόλος των κυνηγών μπορεί να είναι θετικός αλλά και ε, αρνητικός. Πρέπει να εξηγήσει κανείς στους κυνηγούς τι πρέπει να κάνουν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό καταφέραμε στην τσεχική δημοκρατία και γι' αυτό συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Απλώς να συμπληρώσω ότι έχουμε μια στρατηγική διαχείριση των αγριόχειρων, μια ε, στρατηγική σε βάθος χρόνου, η οποία είναι πολύ διεξοδική ε, και σε κάποιες επιτυχίες της ενδεχομένως να μην εκ πρώτης όψεως ακούγεται λογική. Δηλαδή ε, οι κυνηγοί εκ πρώτης όψεως μερικές φορές δεν αντιλαμβάνονται το τι ακριβώς το ζητάμε και το ποια συμπεριφορά είναι λανθασμένη. Ε, για παράδειγμα είναι πολύ ενδεικτικό το παράδειγμα της Τσεχίας. Δηλαδή σε περιοχές όπου ε, όπου υπάρχει ακριβώς η ασθένεια, δεν θα πρέπει να σκοτώνουμε τους αγριόχινους, θα πρέπει να τους αφήνουμε να πεθαίνουν από την ασθένεια. Γιατί αν αρχίσουμε να τους αναρτώνουμε μαζικά, δηλαδή αν εφαρμόσουμε την τεχνική καλάσνικο φως, την ονομάζαμε στη Ρωσία, τότε μπορεί να υπάρχει καταστροφή πραγματικά. Όταν λοιπόν ε, ε, οι κυνηγοί στην αρχή άκουγαν ε, τη ε, ρωσική τηλεόραση και τα όσα ανέφερε, άρχισαν να εφαρμόσουν αυτή την τεχνική Καλάσνικο, να θανατώνουν δηλαδή όλου του αγριόχειρου και αυτό επιδίνωσε πολύ την κατάσταση, ειδικότερα στι δύο βορειότερε χώρε τη Βαλτική, όπω είδαμε και στο χάρτη προηγουμένω. Τώρα, αυτό που κάνουν τώρα στην Τσεχία οι κυνηγοί είναι πλήρης πάυση του κυνηγιού στους, ε, στις περιοχές όπου υπάρχει ε, η ασθένεια. Δηλαδή 50 ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα όπου ουσιαστικά πρόκειται δηλαδή μόνο για, ένα, για μια δασική έκταση. Αντί λοιπόν να θανατώνουν τους αγριόχειρους, δεν θανατώνουν λοιπόν σε αυτή την περιοχή του αγριόχειρου, αντιθέτω σε όλε τι περιοχέ γύρω από αυτήν την πληθυσμένη περιοχή θανατώνουν του αγριόχειρου αλλά και ε, μέσω της απαγόρευσης κάθε είδους χορήγησης τροφής στους αγριοχείρους. Και επίσης η θανάτωση γίνεται στοχευμένα των θηλυκών αγριόχειρων ε, στην αναπαραγωγική ηλικία. Πράγμα βέβαια που δεν αρέσει στους ίδιους τους ε, κυνηγούς, αλλά στους οποίους επιβάλλεται να το κάνουν και στους οποίους δίνονται και εκείνατρα μέσω μιας χρηματικής αποζημίωσης για κάθε θηλυκό αγριόχειρο ο οποίος θανατώνεται. Άρα λοιπόν, η πάυση του κυνηγιού στα hot spots, δηλαδή ε, στις περιοχές όπου είχε ε, εντοπιστεί, ενώ, ενώ η θανάτωση στοχευμένη ε, σε περιοχές όπου είναι ελεγχόμενη ακόμα η κατάσταση, όπως σημαίνει αυτή την περίοδο στην Κροατία, είναι καλύτερη στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο, οι κυνηγοί πράγματι έχουν, κινούνται με τον σωστό τρόπο γιατί δεν εξαπλώνεται προς τα δυστικά, προς τις μας ασθένεια. Ε, αλλά υπάρχει μια εξάπλωση, για παράδειγμα, ε, προς Νότο. Βέβαια, εκεί υπάρχει η περίπτωση της Ουκρανίας, ε, δηλαδή ε, εκεί η εξάπλωση λαμβάνει χώρα γιατί καταλαβαίνετε, αν είναι δύσκολο να πείσουμε κάποιου κυνηγού εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζεστε πόσο δύσκολο να είναι, θα είναι να πείσουμε κάποιου κυνηγού ε, κράτο που δεν είναι ε, κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτά πρέπει να πω. Μισό λεπτό ζήτησε το λόγο και πάλι ο κύριο Άγνιο, οπότε δεν ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Δεν σχολιάσετε αυτό που σας είπα. Πόσο σοβαρή είναι η νόσος για τους αγριόχειρους. Αναρώνουν ποτέ όπως τα κουνέλια από τη μειξωμάτωση και αποκαθίσατε τελικά μια ισορροπία. Όχι, η αρρώστια είναι θανατηφόρα και για τους αγριόχειρους και για τους χείρους ελάχιστη είναι η αγριόχειρη, 0,5% θα μπορούσαν να επιζήσουν ίσως. Αλλά η βιβλιογραφία έχει επιβεβαιώσει ότι σχεδόν 100% των ε, ζώων που έχουν προσβληθεί πολύ σύντομα πεθαίνουν σε 2-3 μέρες. Γι' αυτό και ο Δόκτωρ Ναβαριέγκο σας είπε ότι καλύτερα να αφήσουμε ε, την αρρώστια να σκοτώσει τα ζώα στην περιοχή και ε, να αφήσουμε από μόνη της ε, να κάνει τη δουλειά της όσο και να απομακρύνουμε φυσικά τα κουφάρια για να αποτρέψουμε παραμονή του ιού και εξάπλωση ή μετάδοση σε άλλα ζώα. Η απο, απομάκρυση των κουφαριών είναι πολύ σημαντικό για να ε, ελευθερώσουμε τα δάση από τον ιό. Ιδιαίτερα στο βορρά που υπάρχει παγετό στο χειμώνα και όταν το κουφάρι παγώνει ε, το Δεκέμβριο, το χειμώνα, όταν ξεπαγώνει την Άνοιξη, ε, ο ιός εξακολουθεί να είναι παρός και ενεργό και ξέρετε ότι τα, οι αγριόχειροι τρέφονται με αγριόχειρους, οπότε ε, διαιωνίζεται η νόσος από τη στιγμή που παραμείνουν τα κουφάρια και δεν τα απομακρύνουμε. Η κυρία Σραίρα αλλά παρακαλώ πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις ναι, αλλά και οι λύκοι μπορούν να, να φάνε νεκρά Από ό,τι ξέρω, στο δάσος ισχύει αυτό. Επίσης, ε, οι κάτω χώρες ε, είχαν δυστυχώς μεγάλη εμπειρία από την νόσο αυτή και διδαχθήκαμε πολλά από την εμπειρία μας. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε λοιπόν τις πληγήσεις χώρες να αναπτύξουν μέτρα αντιμετώπισης της ζωονόσου. Σε εμά χρειάστηκε να θανατωθούν εκατομμύρια ζώα, κάτι που ήταν τραγικό για τους κτηνοτρόφους, αλλά την κρίση την ξεπεράσαμε και μπορούμε ε, να βοηθήσουμε με την πείρα μας ε, τις χώρες που αντιμετωπίζουν τώρα το πρόβλημα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γνώση αυτών των πρακτικών και των μέτρων. Ναι. Στις κάτω χώρες είχαμε εδώ αλλά όχι από την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, από την κλασική Πανόλη των Χείρων ε, στα τέλη του 1990 ε, πράγματι 11 εκατομμύρια χείρι τελικά έχασαν πέθανε ε, από αυτή την ασθένεια βέβαια η Αφρικανική Πανόλη των Χείρων συμπεριφέρεται τόσο διαφορετικά από την κλασική Πανόλη ε, είναι δηλαδή πολύ πιο σημαντική ε, για τη μετάδοση της αφρικανικής επανόλης ε, ο αγριόχειρος. Είναι πολύ πιο σημαντικός. Και κατά την παρουσίασή μου είπα ότι ακριβώς λόγω αυτού του κρούσματος στη Ρουμανία και στην Τσεχία είναι σημαντικό για όλα τα κράτη-μέλη, όχι για τις, για τις το να αντιληφθούν ότι ό,τι συνέβη λοιπόν στη Ρουμανία και στη Τσεχία μπορεί να συμβεί και στα ίδια και γι' αυτό ε, έχουν ενταθεί οι εκστρατείε ενημέρωση του κοινού. Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει διανύμει φυλάδια ε, στου οδηγού ε, των φορτηγών που έρχονται από τι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη και υπάρχουν και άλλε δράσει που έχουν λάβει μια σειρά από χώρε και τι οποίε συγχρηματοδοτούμε προκειμένου να μην περάσει στον πληθυσμό των αγριόχειρων αυτών των χωρών η ασθένεια, αλλά ε, και να μην υπάρξει εξάπλωση από τις εκμεταλλεύσεις της χώρας η οι οποίε έχουν πληγεί. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν άλλε ερωτήσει. οπότε ευχαριστώ θερμά τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση. Ακούσαμε πολλέ απορίες και παρατηρήσει. Σήμερα έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου, οπότε δεν χρειάστηκε να περιορίσουμε το χρόνο της συζήτησης ούτε των καλεσμένων, ούτε των ευρωβουλευτών. Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλό βράδυ σε προσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 15, παρουσίαση της έκθεσης από την αποστολή στην Κροατία 19 με 21 Σεπτεμβρίου. Μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας επισκέφθηκε την Κροατία 19 με 21 Σεπτεμβρίου ε, με στόχο να ενημερωθούμε για την πρόοδο που επιτελέστηκε αλλά και για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γερικός κλάδος της Κροατίας. Ε, διαβάζοντας, ε, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα αποτελέσματα της κοινή γεωρικής πολιτικής στην Κροατία από την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου του 2013. Η αντιπροσωπεία οργανώθηκε από τους Κροάτες συναδέλφους μας, την κυρία Μαριάννα Πετήρ και τον κύριο Ιβάν Γιακόφτσιτς, που συνόδευσαν και την αποστολή αυτή, σε συνεργασία με τη γραμματεία της Επιτροπής μας. Στην αντιπροσωπεία αυτή συμμετείχαν ο κύριος Δέση, η κυρία Μίλλερ, η κυρία Σένερα Ροντρίγκες, ο κύριος Μπόγκοβιτς, ο κύριος Ταραμπέλα, ο κύριος Καπούτο και η κυρία Γκοσεύσκα και ο υποφαινόμενος. Είχαμε πολύ εντατικό και πλούσιο πρόγραμμα που μας επέτρεψε να εξοικειωθούμε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην χώρα αυτή, την Κροατία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και πάλι την κυρία Πετήρ και τον κύριο Γιακόφτσιτς για την άρτη οργάνωση. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Πετήρ, κατόπιν στον κύριο Γιακόφτσιτς. Πάντως ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα των επισκέψεων, πολύ ενδιαφέρον το κλίμα μεταξύ μας ε, πολύ θερμό, η προετοιμασία άρτια και η φιλοξενία επίσης θερμή. Πολύ εγκάρδια ατμόσφαιρα επικράτησε και σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύ καλή αυτή οργάνωση της αποστολής μας μια και το πρώτο τμήμα τη ε, αντιπροσωπεία του οργάνωση η κυρία Πετήρ και το δεύτερο ο κύριο Γιακόφτη. Με αυτή τη σειρά να μιλήσουν και οι δύο συνάδελφοι. κυρία Πετήρ, σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και του συναδέλφου που έλαβαν μέρο ε, στην ε, αποστολή αυτή και μπόρεσαν να συναντηθούν επί τόπου με τους παραγωγούς μας στους πιο ευαίσθητους κλάδους γεωργίας, όπως το τομέα προκυπευτικών, το γαλακτοκομικό και τον τομέα παραγωγής χειρίου, και χειροτροφία. Είχαμε επίσης συναντήσεις με νέους γεωργούς, με αμπελουργούς, Κροάτες ε, για ένα τομέα που αποτελεί σημαντικό δυναμικό και ε, αναπτύσσεται σημαντικά. Επίσης, ε, είδαμε τις διαφορές στην ΚΑΠ μεταξύ των παλιών και νέων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το, τη διαφορά συνθήκων μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Είναι σημαντικό λοιπόν από τις συζητήσεις αυτές να λάβουμε υπόψη τα σχόλια των Γεωργών ε, για να διορθώσουμε κάποιες αδικίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην κοινή γεωργική πολιτική γιατί έχουμε κατακλειστεί από εισαγόμενα προϊόντα και μάλιστα που είναι χειρότερη ποιότητα από τα αντίστοιχα προϊόντα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίση να καταπολεμήσουμε τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ. Για μα αυτό είναι προτεραιότητα. Αλλά προτεραιότητα είναι όχι μόνο τη Κροατία αλλά και τη Επιτροπή μα να καταπολεμηθούν αυτέ οι εμπορικέ πρακτικέ. Επίση, κατά ένα πέπτο μειώθηκε η παραγωγή ε, και ε, ενώ σε άλλες χώρες έχει αυξηθεί, έχει διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί η γαλακτοπαραγωγή. Κάτι που δείχνει μεγάλη ανισορροπία και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Επίσης, ε, είναι σημαντικό που μιλήσαμε και με χειροτρόφους γιατί είναι γεγονός ότι ακόμη δεν έχουμε εξασφαλίσει αυτάρκεια στην παραγωγή χείριου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα έχουν τεράστιες ζημιές οι χειροτρόφοι, διπλάσιες σε σχέση με το 2015, ε, ενώ στα σούπερ μάρκετ καταφθάνει κρέας κατεψυγμένο χρόνια ολόκληρα και μετά την απόψυξη γίνεται συσκευασία, ενώ στις ε, ετικέτες δεν αναφέρεται η ημερομηνία της φαγής, γιατί επαναλαμβάνω πρόκειται για κρέας που είναι, έμεινε κατεψυγμένο χρόνια ολόκληρα και αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο. Επίσης, ε, σας ε, δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμάσετε και ένα παραδοσιακό προϊόν που τη χάνει και ονομασίας προέλευσης και μάλιστα έχουμε στενή συνεργασία και με τις αρμόδιες αρχές ώστε αυτό το, το προϊόν να το προωθήσουμε ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Ένα θετικό παράδειγμα ήταν αυτό των ε, βιολογικών μας ε, παραγωγών, βιολογικών γεωργών και νέων γεωργών στην Κροατία. Βέβαια αυτοί επισήμαναν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την πρόσβασή τους στα δάνεια. Ακούσαμε από ε, Γερμανούς συναδέλφους ότι τα επιτόκια στη Γερμανία είναι 0,2%, ενώ στην Κροατία τα επιτόκια είναι 8 με 9% με τόσο υψηλά επιτόκια φυσικά δεν μπορούν οι γεωργοί μας ούτε οι υπόλοιποι Κροάτες να είναι ανταγωνιστικοί. Επίσης, ε, η παραγωγή απορροκυπευτικών παραπονέθηκαν για ε, εισαγωγές απορροκυπευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες ε, ε, που έχουν ε, ε, λάβει φυτοφάρμακα που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δημιουργεί θέμα του ανταγωνισμού. Εμείς ενισχύουμε τους ελέγχους και παρόλα αυτά εισάγουμε προϊόντα που καταπατούν τα δικά μας μέτρα. Αυτό είναι λάθος, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές μας που έχουν δικαίωμα σε υγιεινά και ποιοτικά τρόφιμα και ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατεύσουμε και τους παραγωγούς μας. Επίσης, πολύ επισήμαν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα, αποθεματικό για τις κρίσεις, εκτός του γεωργικού προϋπολογισμού. Αυτό πιστεύουμε και υποστηρίζουμε και εμείς την Επιτροπή Γεωργίου μας. Θέλουμε τέτοιο ταμείο ή αποθεματικό για τις κρίσεις, εκτός του γεωργικού προϋπολογισμού, γιατί μέχρι στιγμής ο γεωργικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των γεωργών μας και άρα δεν μπορεί να καλύψει και τις κρίσεις. Συναντηθήκαμε και με τον Υπουργό Γεωργίας ε, και με τους ε, Προέδρους Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Γεωργίας και ε, Ευρωπαϊκών Επιθέσεων και μάλιστα μεταβιβάσαμε στον Υπουργό μας κάποιες ιδέες της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης είχαμε συναντήσεις και με τομείς ε, αριστείας ε, από τη Γεωργία, με θύλακες ε, τομείς νης στην Κροατική Γεωργία. Αυτή ήταν η τελευταία μας συνάντηση στο Ζάγκρεπ. Ελπίζω με όλες τις εντυπώσεις αυτές που συγκεντρώσατε από την Κροατία θα συμβάλλετε σε συνεργασία μαζί μας για να εξασφαλίσουμε καλύτερες και πιο ποιοτικέ συνθήκε για την Κροατική Γεωργία και την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ο κύριος Γιακόφτσης, ευχαριστώ. Ε, λίγα λόγια θα προσθέσω κι εγώ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που αποφασίσατε να πραγματοποιήσετε αυτή την αποστολή στην Κροατία και σας ευχαριστώ που ήρθατε μέχρι την Ίστρια, την ε, περιοχή στην οποία ήμουν περιφερειάρχης για 20 περίπου χρόνια ε, και που πολύ σοβαρά ασχολούμαστε με την γεωργία, κυρίως την αμπελουργία, την παραγωγή ίνου αλλά και με τη μεταποίηση κρέατος και την παραγωγή γάλακτος, αλλά έχουμε και άλλα προϊόντα, έχουμε αναπτυγμένη γεωργία στην Ιστρία. Επίσης, τονίσαμε την συνέργεια που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ γεωργίας και τουρισμού. Τα προϊόντα της Ιστρίας ε, είναι σχεδόν όλα εξαιρετικής ποιότητας. Το ελαιόλαδο από την Ιστρία είναι ίσως ε, ε, πλήρη της καλύτερες παγκοσμίες προδιαγραφές και μάλιστα φέτος και πάλι η Ίστρια αναδείχθηκε ως η καλύτερη ελαιοπαραγωγός περιοχή του κόσμου. Και από τα 100 καλύτερα δείγματα, 75 ε, ήταν από την Ίστρια, πέραν των δειγμάτων της Ανταλουσίας και της Τοσκάνης. Οπότε ε, έχουμε κορυφαία θέση στην ε, παγκόσμια ελοπαραγωγή. Το θέμα είναι να τη διαφυλάξουμε και να δώσουμε κίνητρα στους παραγωγούς μας και στους γεωργούς μας που ήδη βρίσκονται στην κορυφή να διατηρήσουν τη θέση τους. Θα πρέπει να τροφοδοτήσουμε λοιπόν αυτή την ανταγωνιστικότητα και αυτά τα επιχειρούμε και εντός της ε, Κροατίας, αλλά μια και έχουμε και ευρωπαϊκά κονδύλια, θα πρέπει να φροντίσουμε να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ των διαφόρων περιοχών, γιατί η ε, Τεριέστη που είναι πολύ ανεπτυγμένη δεν μπορεί να πάρει ε, κονδύλια και επίσης ε, δεν θα πρέπει να θέσουμε σε δυσμενή μεταχείριση τις ανεπτυγμένες περιφέρειες γιατί οι ανεπτυγμένες περιφέρειες της Κροατίας δεν είναι εξίσου ανεπτυγμένες οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες περιφέρειες των άλλων χωρών. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και αυτές τις περιφέρειες για να διατηρήσουν την υψηλή θέση και την ποιοτική παραγωγή που έχουν επιτύχει. Σας ευχαριστώ και πάλι για την αποστολή, για την, αποστολή, για την παρουσία σας στην πατρίδα μου. Νομίζω ότι όλοι ε, ικανοποιήθηκαν με την επίσκεψη αυτή. Ακόμη και σήμερα μου στέλνουν ευχαριστήριες επιστολές για την πραγματοποίηση αυτής της αντιπροσωπείας. Σας τις μεταφέρω και ελπίζω να δοθεί μια συνέχεια και να ακολουθήσει και άλλη αποστολή. Να προσθέσω και εγώ καμιά δυο φράσεις, μια και προείδρευσα στην αποστολή αυτή στην Κροατία και να απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις. Όντως υπάρχουν διαφορές στη, και στην Κροατία και εντός Κροατίας ε, ό,τι αφορά το επίπεδο ανάπτυξης των περιφερειών. Και είναι διαφορετικές συνθήκες, ε, διαφορετικό το δυναμικό και διαφορετικές οι ευκαιρίες εντός της Κροατίας. Οπότε στο μέλλον και στη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τέτοιες ιδιαιτερότητες όπως αυτή της Κροατίας και της διαφοράς μεταξύ των περιφερειών της θα πρέπει να αντιληφθούμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες και ποιες οι διαφορές ε, στην κατάσταση της γεωργίας εντός της ίδιας χώρας. Ε, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους ε, των περιφερειών, των τοπικών κοινοτήτων, με τον Υπουργό Γεωργίας στην Βουλή ε, και μάλιστα η κυρία Πετήρ βλέπω ότι έχει άμεσες επαφές ε, και με τους γεωργούς και με τους ε, οικολόγους. Και μάλιστα όταν περούσαμε από τις διάφορες πόλεις βλέπω ότι υποκλίνονταν μπροστά στην κυρία Πετήρ, τη χαιρετούσαμε ιδιαίτερο σεβασμό. Και εγώ κατάλαβα πως ε, προσπαθούμε να αφιερώσουμε κονδύλια και στην υπόλοιπη Κροατία, όπως έγινε και με την Ίστρια. Αλλά γι' αυτό θα περάσει ίσως α, κάποιος χρόνος. Γι' αυτό είναι σημαντικό που οι Κροάτες Ευρωβουλευτές στηρίζουν ιδιαίτερα τις περιφέρειες αυτές, αλλά και την ανάπτυξη του περιβάλλοντος στην Κροατία. το πρώτο τμήμα της αντιπροσωπείας ήταν ίσως πιο έντονο. Εγώ δεν το ένιωσα ότι ήταν παραφορτωμένο το πρόγραμμα, ίσως γιατί καθυστέρησα, δεν έφτασα από την αρχή. Πάντως ήταν πολύ ενδιαφέρουσε όλες τις συναντήσεις που είχαμε με προσώπους των διαφόρων κλάδων. Και άκουσα τη στρατηγική και από αυτή διαβλέπω και το μέλλον της Κροατίας. Βλέπω ότι έχετε ε, πολύ καλή εστίαση και όραμα για την ανάπτυξη. και ήταν τόσο θετικές οι εντυπώσεις μας που σίγουρα πολύ θα επιστρέψουμε και για διακοπές στην Κροατία. Πάντως είναι, ήταν πολύ σημαντική η αποστολή μας. Επιβεβαιώνω την ποιότητα του ελαιολάδου και του ίνου δεν είναι ανταγωνιστικά αυτά τα προϊόντα. Σε χαρητήρια. Και πιστεύω ότι και εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε σχέσεις και επαφές με τους συνομιλητές μας και στην Κροατία. Ευχαριστώ κυρία Γκιλέρα. Ναι, δυστυχώς εγώ δεν είχα την ευκαιρία να πάω στην Κροατία, αλλά τη γνωρίζω και για λόγους τουριστικούς και για λόγους... Ναι, στο μέλλον θα πάτε. Ούτως ή άλλως εγώ είμαι και από χώρα με υψηλό τουρισμό όπως ε, η Ισπανία, αλλά ξέρω την Κροατία και για λόγους εργασίας. Θα ήθελα να γνωρίσω την ε, ε, προσπάθεια των συναδέλφων, την εργασία τους, γιατί γνωρίζω ότι κάνουν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου στην Ίστρια κάνουν εξαιρετική εργασία και το λέω γιατί εγώ Προέρχομαι από περιφέρεια ελαιοπαραγωγό που ξέρει εδώ και αιώνες ε, να καλλιεργεί το ελαιόλαδο, να παράγει το ελαιόλαδο και μπορώ να, ε, ε, δεν μπορώ παρά να εγκομιάσω ακριβώς αυτήν την προσπάθειά τους. Ε, και τα προβλήματα των γεωργών στην ε, Κροατία είναι παρόμοια με τα προβλήματα των άλλων γεωργών. Ωστόσο, η προσπάθεια που καταβάλουν ε, και αυτή η προσπάθεια που κάνουν να συνδέσουν το γεωργικό προϊόν με το τουριστικό προϊόν είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, όπως είπε και η κυρία Πετήρ, αλλά ε, σίγουρα στο μέλλον ε, θα έχουν πολύ καλές εξελίξεις γιατί σας είπα ξέρω τη δουλειά που κάνουν ε, για το ελαιόλαδο και εγώ που έρχομαι από την Ανδαλουσία μπορώ να αναγνωρίσω την καλή δουλειά που γίνεται για αυτό το τομέα. Ξέρω ότι ακριβώς επειδή είστε ειδήμος σε θέματα ελαιολάδου οι δικές σας κρίσεις αξιολογικές για τέτοια θέματα είναι πολύ έγκυρες και αξιόπιστες. Άλλος κανεί θέλει το λόγο? Όχι. Οπότε θα ήθελα και πάλι θερμότατα να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Γιακόφτσιτς και την κυρία Πετήρ για την άρτια οργάνωση. Θα θυμόμαστε ε, συνεχώς αυτή την πολύ καλή ατμόσφαιρα που ήταν και θερμή και φιλόξενη αλλά και μεστή ε, αυτό το πρόγραμμα με πολλές συναντήσεις. Θα το θυμάμαι όσο ζω λοιπόν. Ήταν πολύ ευχάριστη εμπειρία. Θερμά ευχαριστώ λοιπόν για όλη τη δουλειά και την προσπάθεια και μία παρατήρηση μου έμεινε. Δεν βλέπω σε αυτό το ωραίο φυλάδιο το ταπεινό μου πρόσωπο. Τι, δεν είμαι και τόσο μικρό όμω για να περάσω απαρατήρητο. Μήπως επειδή άργησα, με τιμωρήσατε και δεν με περιλάβατε στο έγγραφο αυτό, φυλάδιο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πέραμε στο τελευταίο σημείο, επιβεβαίωση των αποφάσεων των συντονιστών. Σα στείλαμε ηλεκτρονικά τις αποφάσεις των συντονιστών, αλλά και εγγράφος. Έχετε λάβει το σχετικό κείμενο. Διάφορα υπάρχουν παρακαλώ. Όχι. Οπότε επόμενη συνάντηση αύριο. Αύριο σε 9. Κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Παρακαλώ δώστε το παρόν να μην είναι μόνο ε, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Εγώ δυστυχώ κολλείω με αύριο, φεύγω ταξίδι, θα με αντικαταστήσει ο κύριος Δεκάστρο. Επόμενη συναντήση 6 Νοεμβρίου, 9 Νοεμβρίου, 22 και 23 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Θα σας στείλουμε ενημέρωση πιο διεξοδικά. Σας ευχαριστώ και πάλι τους επισκέπτες μας, τους διερμηνείς, τη γραμματεία. Καλό σας βράδυ. Ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα και νωρίτερα τελειώσαμε και ταυτόχρονα δεν περιορίσαμε κανένα στο χρόνο αγόρευσης. Πολύ ωραία. Καλό σας βράδυ.